knows uh, Συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, παρακαλώ καθίστε. Καλησπέρα σε όλους. Συγχαρητήρια και πάλι ευχές μάλλον προς τους Ρουμάνους συναδέλφους και των δύο επιτροπών. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν υπάρχουν σχόλια, εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη χωρίς αλλαγές. Δεν βλέπω να θέλει κανείς να σχολιάσει. Ανακοινώσεις. Δύο ανακοινώσεις. Η συνεδρία μεταδίδεται στο διαδίκτυο. Και δεύτερον έχουμε διερμηνία σε 22 γλώσσες. Ως ήθιστε, γνωρίζετε πολύ καλά ποια διαδικασία επιβάλλεται για τις κοινέ συνεδριάσεις. Σας καλωσορίζω όλους. Μαζί συντάσσουμε αυτή την σημαντική έκθεση. Έχουμε προβλέψει δύο ώρες για αυτή τη συζήτηση. Και από τις προηγούμενες συνεδριάσεις προέκυψε συμφωνία μεταξύ των δύο επιτροπών σε κάθε κοινή συνεδρία συνεπάρχει συμπροεδρία των δύο προέδρων, της κυρίας Βίκη Φόρντ και ε, μου του ιδίου. Έχουμε 1287 τροπολογίες, χωρίς να μετράμε τις νομοδοτήσεις των υπολείπων επιτροπών. Έχουμε όλες τις νομοδοτήσεις μπροστά μας και πραγματικά να συγχαρώ και τους δύο συνεισηγητές πρώτα την κυρία Κέπχαρτ και την κυρία Κάλλας. Εξαιρετική δουλειά. Και φανταζόμαστε ότι δεν είναι απλό να συνεργαστείτε με τόσους πολλούς σκιώδεις εισηγητές ταυτόχρονα. Συγχαρητήρια λοιπόν και σε όλους τους σκιώδεις, από όλες τις επιτροπές και από τις δύο επιτροπές. 15, 16, 17 άτομα Και δεν μετράω καν τους συνεργάτες, τους υπευθύνου της γραμματείας, των οποίων η συνδρομή είναι πολύτιμη. Ο σκοπός της σημερινής ανταλλαγής απόψεων είναι να δούμε τις πολλαπλές συμβαστικές τροπολογίες για τις ε, πολλές παραγράφους που μας απασχολούν, αλλά έχουμε συμφωνήσει με την κυρία Βεκιφόρντ. Οι δύο εισηγητριές μας και οι σκιώδεις να μας πούν όσο μπορούν περισσότερα. Και για τα άλλα σημεία, τι συμβαστικέ τροπολογίε που ενδεχομένως τις αποσχολούν, που δεν έχουν ολοκληρωθεί απαραίτητος, ίσως να είναι ακόμη σημαντικότερα από την ε, οπτική γωνία της δικής μας συζήτηση. Διότι αν έχετε λάβει συμβαστική πρόταση για 10-12, δεν έχει σημασία πόσες τροπολογίες, το θέμα είναι τι γίνεται και με τα υπόλοιπα. Αυτό είναι το σημαντικότερο ίσως. Εάν μπορείτε λοιπόν να μας παρουσιάσετε τη θέση σας. Το ίδιο και σκιώδης. Παρακαλώ εξηγήστε μας τις απόψεις σας. Θα συμπεριλάβουμε βεβαίω δι και τις υπόλοιπες νομοδοτήσεις και στον κατάλογο ψηφοφορίας, τις συμβαστικές τροπολογίες των υπολείπων επιτροπών. Είμαστε λοιπόν στην αρχή της συζήτησής μας. Έγκριση των πρακτικών της, προηγούμενη της προηγούμενης συνεδρίασης, τα οποία περιλαμβάνονται στους φακέλους των βουλευτών από τη συνεδρία της 10 Νοεμβρίου 2015. Εάν δεν υπάρχουν άλλα σχόλια, θεωρούμε ότι έχουν εγκριθεί τα πρακτικά, δεν υπάρχουν σχόλια. Και τώρα να ζητήσω τη συμπρόεδρο, την κυρία Φόρντ, να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ, συμπρόεδρε. Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε σήμερα. Απλώς να αποσαφηνίσω ακριβώς που έχουμε φτάσει. Θέλουμε να ψηφίσουμε το κυβερνητικό ψήφισμα στις 14 Δεκεμβρίου. Γνωρίζουμε ότι η Επιτροπή σκοπεύει να υποβάλει προτάσεις την ερχόμενη εβδομάδα Οπότε θα ήταν πολύ καλό σε αυτή μας τη συζήτηση όχι απλώς να συζητήσουμε τις συμβαστικές προτάσεις εκ των οποίων υπάρχει συμφωνία, αλλά να συζητήσουμε και αυτές που είναι αμφιλεγόμενες. Έτσι θα διευκολύνουμε και τι τις μα μας και τους συζητητές και εάν οι βουλευτές έχουν συγκεκριμένες προτάσεις, συγκεκριμένα σχόλια για τις προτάσεις που μπορεί να ανακύψουν την ερχόμενη εβδομάδα, Ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ακούει προσεκτικά, διότι το Κοινοβούλιο μπορεί να αποκλίνει κάπως από την ε, τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς αυτά που σκοπεύουν να αναγγείλουν την ερχόμενη εβδομάδα. Ελπίζω λοιπόν να μας ακούσετε και αυτή θα είναι η τελευταία ευκαιρία που θα έχουμε να ε, αφουγκραστούμε και να αξιοποιήσουμε τη συλλογιστική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μπούζεκ, ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Τρεις εβδομάδε λίγο πολύ για να περατώσουν τις εργασίες μας. Δεν μένει λοιπόν πολύς χρόνος. Θα ξεκινήσω από τις συνεισηγήτριες. Έχετε συμφωνήσει ποια θα λάβει το λόγο πρώτη. Έτσι φανταζόμουν ότι τα έχετε κανονίσει μεταξύ σα. Κυρία Γκέπχαρτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το κάνουμε εκ περιτροπής. Προχωρούν λοιπόν οι εργασίες μας. Δεν είναι πάντα πολύ απλό, αυτό είναι σωστό, γιατί υπάρχουν διαφορετικές απόψεις μεταξύ των πολιτικών ομάδων και εν μέρη πρέπει να περιμένουμε και τις ε, γνωμοδοτήσεις ε, των επιτροπών που πρέπει να γνωμοδοτήσουν, διότι με βάση το άρθρο 54 πρέπει να λάβουμε υπόψη τα θέματα αρμοδιότητάς τους. Αυτή τη στιγμή εκπονούμε 38 συμβαστικές τροπολογίες σε τέσσερα τμήματα. Τα δύο πρώτα ε, σύνολα τροπολογιών είναι σχεδόν έτοιμα Χρειαζόμαστε λίγες συζητήσεις ακόμη, αλλά μπορούμε να πούμε ότι στην ουσία έχουν κλείσει οι συζητήσεις. Τα δύο επόμενα τμήματα τροπολογιών ήδη τα συζητάμε και εν μέρη έχουμε καταλήξει με τους ε, σκιώδεις και τους ε, συντάκτες γνωμοδοτήσεων έχουμε καταλήξει σε κάποιες διατυπώσεις και την επόμενη πέμπτη, την ε, προσεχή πέμπτη δηλαδή μεθαύριο θα προχωρήσουμε. Βέβαια δεν μπορώ να σας παρουσιάσω τώρα όλες και τις 38 τροπολογίες, οπότε θα ακολουθήσω τη συμβουλή σας. Θα σας πω ποια θέματα είναι πολιτικά πιο συζητήσιμα, γιατί υπάρχουν ακόμη ανταλλαγές ε, απόψεων και για αυτές ακριβώς τις τροπολογίες είναι και πιο δύσκολο να καταλήξουμε στη συμφωνία. Αρχίζουμε την παράγραφο 15 για την παράδοση πακέτων ταχυδρομικών δεμάτων. Ε, το θέμα είναι πόσο ευρέως πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Όλοι συμφωνούμε ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα για τις ε, διασυνοριακές ε, δοσοληψίες ε, ηλεκτρονικού εμπορίου. Πρέπει να δούμε και το κόστος που προκύπτει, την ταχύτητα με την οποία ε, παραδίδονται, αλλά και την ασφάλεια των, παρα, ε, προϊόντων. Θεωρώ ότι από την έμπλα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι το θέμα δεν είναι μόνο η τιμή, αλλά και επιπτώσεις ε, για τον κόσμο της εργασίας, τους εργαζόμενους, και την ποιότητα της δουλειάς τους. Πρέπει να ληφθεί υπόψη και αυτό. Αυτό είναι ένα θέμα που το συζητάμε μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Η άποψή μου είναι ότι η Επιτροπή Απασχόλησης έκανε μια πολύ καλή πρόταση, την οποία θα μπορούσα να δεχθώ. Είναι λίγο πιο ήπια από αυτά που έχω υποβάλει εγώ μέσω των τροπολογιών μου, αλλά θα μπορούσε να είναι μια καλή βάση συμβιβασμού. Επίσης είχαμε πολλές συζητήσεις, έντονες συζητήσεις για τις πλατφόρμες και τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Και η κυρία Καλάς και εγώ είχαμε ε, υποβάλει στους ε, σκιώδεις διαφορετικές προτάσεις συμβιβασμών γιατί δεν μπορούσαμε να συμφωνήσουμε, αλλά μεταξύ έχει προχωρήσει η συζήτηση, ούτω ώστε να μπορώ να πω ότι έχουμε μια κοινή συζήτηση, μια κοινή συγγνώμη, υποβολή τροπολογιών. Θέλουμε να κάνουμε μια σαφή διαφοροποίηση μεταξύ μιας πλατφόρμας ως ε, δομής και του τρόπου λειτουργίας, του τρόπου αξιοποίησης της και από την άλλη μεριά τις υπηρεσίες που θα παρέχονται μέσω της πλατφόρμας αυτής. Νομίζω ότι επιτύχαμε μέσω της συζήτησης να συμφωνήσουμε σε αυτήν τη διαφοροποίηση. Γιατί ένα πρέπει να είναι απόλυτα σαφές. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε όλα στο ίδιο σακί. Οι πλατφόρμες και ο τρόπος λειτουργίας τους είναι διαφορετικές μπορούμε να πούμε κάτι για τη δομή τους, αλλά πέρα από τη δομή τους ε, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα περισσότερο. Οι υπηρεσίες που παρέχουν είναι τόσο διαφορετικές που δεν είναι δυνατόν να καταλήξουμε σε ενιαίους ορισμούς. Υπάρχουν πολλές τροπολογίες ε, που επιδιώκουμε αλλά που επιδιώκουν ορισμένοι, αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να φύγουμε προς όλες τις ε, κατευθύνσεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, τι μπορεί να προσφέρει το ηλεκτρονικό εμπόριο, δωμάτια ξενοδοχείων ε, από τη μία μεριά ή ε, ταξί. Από την άλλη μεριά υπάρχουν πλατφόρμες οι οποίες προσφέρουν επιστημονικές υπηρεσίες. Δεν μπορούμε όλα να τα βάλουμε στην ίδια κατσαρόλα, οπότε είναι καλό να υπάρχει διαφοροποίηση. Και για τις πλατφόρμες υπηρεσιών. Τίθεται το θέμα πόσο ολιστικά θα το προσεγγίσουμε. Η ΙΜΚΟ έχει παραδοσιακά εδώ και πολλά χρόνια για τα θέματα αυτά ε, έχει την ε, παράδοση λοιπόν να λέει ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε μεμονωμένα τις ε, υπηρεσίες πρέπει να το αντιμετωπίζουμε σφαιρικά δηλαδή και τις υπηρεσίες και τις επιχειρήσεις ανάλογα αν είναι μικρομεσαίες ή μεγάλες αλλά και τους εργαζόμενους δηλαδή να αναφερθούμε σε όλα τα προβλήματα αυτή είναι μία από τις ιδιαίτερες δυσχέρειες που έχουμε, αλλά νομίζω ότι παρόλα αυτά έχει υπάρξει μία προσέγγιση, ένα συγκερασμός απόψε. Πρόεδρος, με συγχωρείτε. Κοιτάξτε, ε, βλέπετε τι χρόνος προβλέπετε μπροστά σας. Επειδή όμως είναι πολύ περίπλοκο το θέμα, έχετε άλλα δυόμιση λεπτά, συνολικά εννέα λεπτά η κάθε εισηγήτρια. Αλλά όχι περισσότερο παρακαλώ συνεχίζει ο πρόεδρος διότι η κυρία Γκέπχαρντ. Ναι, ναι, εσείς μου ζητήσατε να σας πω πού είναι τα προβλήματα, σε ποιου τομείς, σε ποια σημεία για να βρούμε τροπολογίες. Αλλά παρόλα αυτά έχουμε προχωρήσει αρκετά. Υπάρχουν άλλα θέματα που πρέπει να συζητήσουμε. ή τηλεπικοινωνίες. Αυτά θα τα παρουσιάσει περισσότερο η κυρία Κάλλας, γιατί είναι περισσότερο αρμοδιότητα ήτρε. Επίσης, τίθενται τα θέματα της κυβερνοασφάλειας, παρανόμου περιεχομένου στο ίντερνετ. Δεν τα έχουμε συζητήσει ακόμη αυτά, γιατί πρέπει να τα δούμε και με τη ΛΥΜΠΕ. Και κατά λίγο, κατά τουλάχιστον αυτή την πρώτη παρουσίαση, ίσως να χρειαστεί να επανέλθω αργότερα. Κατά λοιπόν, με το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων γιατί μαζορίζει κάπως αυτό το θέμα και σχετίζεται και με αρμοδιότητες Κουλτ και Γιούρι. Αλλά και από αυτό νομίζω ότι έχουμε προχωρήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Κάλλας. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συνεισηγητές και τους κοιόδης εισηγητές ε, για την πολύ καλή συνεργασία, όπως επίσης και τους βοηθούς και τους συμβούλους, ε, γιατί πολλή δουλειά έχει γίνει για την έκθεση αυτή. Όσον αφορά τα γενικά ζητήματα, θα ήθελα επίσης και, και εγώ να πω ότι η δομή της έκθεσης ε, μας υπευλήθη από την Γραμματεία. Είναι καλό ότι την ε, τηρήσαμε και μάλιστα τηρήθηκε και στις γνωμοδοτήσεις ε, για την ε, δική μας έκθεση. Πρέπει να είμαστε κάπως, να τηρήσουμε κάποια αναλογικότητα δεδομένων και των αποκλειστικών αρμοδιοτήτων κάποιων άλλων επιτροπών. Θα ήθελα και εγώ να ξεκινήσω με τις πλατφόρμες, γιατί αυτό είναι το πιο αμφιλεχόμενο ζήτημα και υπήρξε εκεί η περισσότερη συζήτηση και μάλιστα εκρεμεί και συμβιβασμός ε, επί των ε, πλατφορμών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει αυτή η φιλική προς την καινοτομία για τις πλατφόρμες, κάτι το οποίο θα παροτρύνει ε, ε, τον ανταγωνισμό και θα διευκολύνει την είσοδο στην αγορά. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να μας βοηθά να καταλάβουμε ποια είναι τα προβλήματα με τις πλατφόρμες ε, και όπως είπε και η κυρία Γκέμπχαρτ, το κατά πόσο δηλαδή το πρόβλημα αφορά την πλατφόρμα ή τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της πλατφόρμας. Πρέπει λοιπόν να είναι πολύ σαφές αυτό και κάτι που είναι επίσης σημαντικό είναι να καταλάβουμε από πού προέρχεται το πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα προερχόμενο από κάποιους ε, τομείς επιχειρηματικούς που προσπαθούν ε, να διατηρήσουν το επιχειρηματικό τους ε, μοντέλο που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν σε απαιτήσει της ψηφιακής αγοράς ή κάποιο άλλο θέμα. Ένα ακόμη ζήτημα είναι η αποτελεσματικότητα. Αυτό που, ήταν πάρα πολύ, που μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ είναι η περιορισμένη ευθύνη των ενδιαμέσων και όπως είχαμε πει, ε, είπαν και πολλοί εμπειρογνώμονες, ε, το να φύγει κανείς από αυτήν την περιορισμένη ευθύνη θα είναι πάρα πολύ δαπανηρό, ειδικότερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μπορεί να ε, είναι καλό για τις μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις, αλλά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν αν δεν υπάρχει ολόκληρη στρατιά νομικών ε, και άλλων ανθρώπων που να μπορούν ε, να ε, τους βοηθήσουν να εφαρμόσουν τους κανόνες. Τελικά θα αναγκαστούν να διακόψουν τη δραστηριότητά τους και αυτό δεν είναι αποφελές για κανένα. Δεν υπάρχει μόνο το οικονομικό αλλά και το κοινωνικό κόστος. Επηρεάζει την ελευθερία της έκφρασης γιατί αν για παράδειγμα οι πλατφόρμες έχουν πλήρη ευθύνη και αρχίζουν για παράδειγμα να κλείνουν ένα περιεχόμενο λόγω κάποιων κινδύνων που μπορούν να, που μπορούν να υπάρχουν, φαντάζεστε τι, θα μπορέσει, τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Τι ακριβώς εννοούμε ε, όσον αφορά τον ανταγωνισμό. Μιλάμε για αθέμητο ανταγωνισμό ή μιλάμε για τη διάκριση μεταξύ των αποτελεσμάτων μιας αναζήτησης. Ε, γιατί πρέπει να δούμε τι εννοούμε με ε, την έννοια διάκριση. Πρέπει να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε αυτήν τη σύγχυση. Η ιδέα είναι να μπορούμε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα με την αναζήτηση. Συνεπώς δεν συμφωνώ με την ουδετερότητα των πλατφορμών, αλλά έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε. Για άλλα θέματα, για παράδειγμα τις τηλεπικοινωνίες, συμφωνούμε όλοι ότι ο ανταγωνισμός είναι καλός και αυτό που πρέπει επίσης να επισημάνουμε είναι ότι είναι πολύ σημαντικό να διατηρηθεί η πρόσβαση στα ε, δίκτυα κανόνες για τους παρόχους υπηρεσιών και από την άλλη ε, πρόσβαση ε, στα δίκτυα προκειμένου να ε, γίνει η παροχή κάποιων υπηρεσιών. Κάτι πολύ σημαντικό για την οικοδόμηση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς είναι η επιβολή. Όταν μιλάμε λοιπόν για έναν αρμονισμένο πλαίσιο, για παράδειγμα πώς θα είναι κατάλληλο για την ψηφιακή εποχή ε, εννοούμε πώς θα λειτουργήσει στην πράξη και όσον αφορά την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο νομίζω ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη ε, τις διαπραγματεύσεις ε, που γίνονται αυτή τη στιγμή όσον αφορά την προστασία των δεδομένων και κάτι που θα ήθελα να τονίσω εν προκειμένου είναι ότι πολλές επιχειρήσεις και πολλοί χρήστες δεν, κάνουν, δεν, δεν παίρνουν τα απαραίτητα μέτρα για να περιορίσουν τη ταυτότητα των χρηστών τους, ε, ε, για παράδειγμα κατά την αναβάθμιση του λογισμικού του τους, ε, για παράδειγμα την κωδικοποίηση, την κρυπτογράφηση των δεδομένων, δεν καταλαβαίνουν τι χρειάζεται να γίνει προκειμένου να παραμείνει η επικοινωνία ασφαλής. Επομένως πρέπει να υπάρξουν ε, λύσεις ε, στον κυβερνοχώρο που να ανταποκρίνονται στις ε, στο πραγματικό κίνδυνο. Χαίρομαι όλος ιδιαίτερος που οι περισσότερες πολιτικές ομάδες επιμένουν στις εξελίξεις που μπορεί να έχει αυτό για, τον, για τους πολίτες μας. Όσον αφορά τώρα την τρίτη παρτίδα συμβιβαστικών τροποπολογιών, δεν, αν δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε μεταξύ μας για κάποια θέματα, ίσως θα έπρεπε τα επίμαχα ζητήματα να προτείνουμε να ψηφιστούν ξεχωριστά αλλά τουλάχιστον να δούμε ποιε είναι οι συμβιβαστικέ τροπολογίες που μπορούν να υποστηρίξουν οι περισσότερε πολιτικές ομάδες και να προχωρήσουμε, ώστε όλοι μας να είμαστε λίγο πολύ ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και τι δύο. Ε, πραγματικά, δίκιο έχετε. Αν είναι, είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να επιτύχουμε έναν ε, συμβιβασμό. Αλλά να μην θυμώσει και κανείς στο τέλος, να μην είναι κανείς δυσαρεστημένος, γιατί ε, ε, Μπορεί να μην μπορούμε να βρούμε μια λύση που να μας αφήσει όλους 100% ικανοποιημένους. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ γιατί ε, τονίσατε τα πιο σημαντικά ζητήματα. Να περάσουμε τώρα στους κοιόδης εισηγητές. Ε, η ομάδα του ΕΛΚ πρώτα, ο Φιλίπ Ζουβάν από την Επιτροπή ΙΜΚΟ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα επικεντρωθώ στο θέμα των πλατφορμών και μόνο στην παρέμβασή μου. Πιστεύω ότι το πρόβλημα εδώ είναι διτό. Κατά πρώτον πρέπει να δούμε την ευθύνη που θα έχουν οι πλατφόρμες και πώς θα καταναμηθεί η αξία, παρόλο που δεν είναι αυτό ακόμα το αντικείμενο της συζήτησης. Ως προς την ευθύνη, η δυσκολία ποια είναι ότι η οδηγία του 2000 για το εμπόριο στο άρθρο 14 μιλά για περιορισμό των ευθυνών ε, στις πλατφόρμες, διότι δημιουργείται ένα νέο οικονομικό μοντέλο. Προκειμένου λοιπόν να μην ε, δυσκολέψουμε την ανάπτυξή τους, δεν δώσαμε καμία ευθύνη στις πλατφόρμες. Σήμερα ποια είναι η συνέπεια ότι η καταπολέμηση του παράτυπου εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών, περιεχομένων μάλλον, παρανόμων περιεχομένων, δεν ε, μπορεί να ελεγχθεί στι πλατφόρμες. Δεν έχουν σαφή υποχρέωση οι πλατφόρμες να μας βοηθήσουν στην καταπολέμηση του παράνομου και παράτυπου εμπορίου. Όμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το γνωρίζετε όλοι και εσείς ε, κύριε Πρόεδρε, υπήρξατε και πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πλούσια γιατί μπορεί ακριβώς να δημιουργεί. Εάν τη δημιουργία δεν την ε, μοιραζόμαστε, δεν θα υπάρχει δημιουργία πλούτου. Πρέπει λοιπόν να ε, συμβάλλουν στην καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας αγαθών οι πλατφόρμες εάν θέλουμε να προχωρήσουμε. Θα μπορούσε να υπάρχει ένα πολύ περίπλοκο σύστημα νομοθετικό με πολλούς κανόνες ή να αφήσουμε την κατάσταση όπως έχει σήμερα, αλλά θα συνεχίσουν να ανθούν ε, οι παράνομες συναλλαγές ε, και θα πρέπει να βρούμε ή να επιλέξουμε την ακραία λύση της ε, του περιορισμού ε, των περιεχομένων. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε μία μέση λύση όπου να υπάρχει και ελεύθερη ροή στις πλατφόρμες αλλά και να έχουμε την κατάλληλη προστασία. Και για την κατανομή της αξίας, παρόλο που ακόμη δεν είναι το θέμα μας, αλλά μια μέρα θα πρέπει να το θίξουμε, θα σας δώσω δύο αριθμούς. Το YouTube με 800 εκατομμύρια χρήστες ε, έχει 640 εκατομμύρια κέρδος ετησίως Ενώ η Deezer έχει ένα διστό χρόνο με πολύ λιγότερους χρήστες. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς ακριβώς θα ρυθμιστεί η σχέση της κατανομής αξίας με τις πλατφόρμες και τον αριθμό χρηστών. Ευχαριστώ. Για τους χιώδεις εισηγητές παρακαλώ όχι πάνω από τρία λεπτά. Σεβαστήκατε πλήρως το χρόνο σας. Η κυρία Βιρκούνεν και πάλι από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, να ευχαριστήσω και τους δύο εισηγητές και τις ομάδες τους για τη σκληρή τους δουλειά. Δεν είναι εύκολη διαδικασία να, συντα... να συντάσει κανείς κοινέ εκθέσεις και κοινέ συμβαστικέ λύσεις. Νομίζω όμως όλες οι ομάδες έδειξαν ιδιαίτερη αφοσίωση για να επεξεργαστούν τις συμβαστικέ λύσεις και να σεβαστούν το πολύ πιεστικό χρονοδιάγραμμα. Νομίζω έχει επιτελεστεί πολύ πρόοδο κατά τι διαπραγματεύσει και πολλέ από τι συμβαστικέ ήδη μπορούν να γίνουν αποδεκτέ από όλε τι ομάδε. Όμω, πολλή δουλειά πρέπει να γίνει ακόμη και πολλά θέματα παραμένουν ανοιχτά. Εκεί θα πρέπει να βρούμε μία λύση τι ερχόμενε ημέρε. Διότι έχουμε μόνο μία εβδομάδα για να βρούμε τι ε, συμβαστικέ λύσει. Υπάρχουν κάποια ζητήματα που είναι πιο περίπλοκα από άλλα. Οι άλλοι εισηγητές, ο συνάδελφος Ζουβά ε, ήδη ανέφερε το θέμα που θέτουν οι πλατφόρμες. Βεβαίως υπάρχει ανάγκη να έχουμε έναν ορισμό των διαφορών ειδών που μπορεί να έχουν οι πλατφόρμες, καθώς και ποιο θα είναι το νομικό τους καθεστώς ε, και οι υποχρεώσεις τους και τι γίνεται με τους παρόχους περιεχομένου. Επίσης πρέπει να δούμε αν υπάρχει ανάγκη για επιπλέον ε, νομοθέτηση ή εάν πρέπει απλώς να εφαρμοστούν οι υπάρχοντες κανόνες και νόμοι. Να δούμε αν είναι αυτή η αν πρεπει απλως να εφαρμοστουν οι υπαρχοντες κανονες και νομοι να δουμε αν ειναι αυτη η λυση Για το ΕΛΚ είναι σημαντικό να δημιουργηθεί μια πολιτική φιλική προς την κοινοτομία που να ε, επιτρέπει την πρόσβαση στην αγορά και, να, και τον δίκαιο ανταγωνισμό. Μια από τις βασικές αρχές στην εκθεσή μας θα μπορούσε να είναι ότι Προσπαθούμε να έχουμε ένα πλαίσιο με τους ίδιους κανόνες για παρόμοιες υπηρεσίες, εφόσον είναι επιγραμμικές ή εφόσον δεν είναι στο διαδίκτυο. Ε, θα πρέπει να καθορίσουμε αυτή την αρχή στην έκθεσή μας. Συνολικά, ένα πράγμα που θα θέλαμε να δηλώνεται ξεκάθαρα στην έκθεση είναι ότι τι κίνητρα θα δώσουμε, γιατί δημιουργούμε την ψηφιακή ενιαία αγορά και γιατί είναι αυτό τόσο σημαντικό. Η ενιαία αγορά στον ψηφιακό χώρο είναι ακρογωνιαίο λίθο για να δημιουργηθούν θέσει εργασία και ανάπτυξη στην Ευρώπη. Γι' αυτό το κάνουμε όλο αυτό το εγχείρημα. Γι' αυτό συντάσσουμε και αυτή την έκθεση. Ξέρουμε ότι η απασχόληση και δουλειέ στην Ευρώπη πρέπει να συμβαδίσουν με τους ρυθμούς άλλων μεγάλων πρωταγωνιστών, όπως είπα και η Κίνα. Το ΕΛΚ λοιπόν έχει σκοπό να εργαστεί σκληρά τις επόμενες ημέρες ε, με συνεργασία όλων των σχεδόν εισαγητών για να υποβάλουμε τις ε, κατάλληλες συμβαστικές λύσεις και να ολοκληρώσουμε γέρος. Πρέπει να υποβάλουμε σύντομα το ψηφιακό μαθηματολόγιο εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολύ γρήγορα θα υποβάλει τις πρώτες τις νομοθετικές προτάσεις τους ερχόμενους μήνες. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να εργαστούμε σκληρά τις ερχόμενες ημέρες για να ψηφίσουμε στο Στρασβούργο όπως έχει προγραμματιστεί. Ευχαριστούμε. Να θυμίσω σε όλους σας, σε όλους σας που ετοιμάζεστε στο δεύτερο γύρο να πάρετε το λόγο μετά τους κοιόδους εισηγητές, η καλύτερη λύση θα ήταν να σηκώσετε από τώρα τα χέρια σας και να ζητήσετε το λόγο για να ετοιμάσουμε, για να τον κατάλογο αγωνιτών. Ο συνάδελφος Ζωρίνιου για τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες και την Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η κυρία Ντανάτο ε, δεν μπορούσε να είναι εδώ σήμερα, ε, γι' αυτό θέλω να τονίσω εγώ τα σημαντικότερα στοιχεία αυτού του θέματο. Είναι πολύ σημαντικό να καλύψουμε το ψηφιακό χάσμα στην Ευρώπη και να αντιμετωπίσουμε τα μονοπόλια. Πρέπει να περάσουμε γρήγορα στα επόμενα δίκτυα 5G και στην ε, ανάπτυξη του διαδικτύου για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Επιπλέον Πρέπει να δούμε την, ε, τις επιπτώσεις της ψηφιοποίησης στην κοινωνία και την παγκόσμια οικονομία. Στις συμβαστικές μας λύσεις Θέλω να τονίσω ότι το ψηφιακό χάσμα ως προς τις υποδομές, την βιωσιμότητα και τις ψηφιακές δεξιότητες ε, μας ε, απασχολεί ιδιαίτερως για να οδεύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, στη σωστή κατεύθυνση στην ψηφιακή συμμετοχή. Θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε κάθε ευκαιρία για να υπάρχει ευρυζωνική πρόσβαση για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες ασχέτως του που ζουν. Ε, σε περιοχές της υπαίθρου ή σε αστικά κέντρα. Τα, οι δεξιότητες του διαδικτύου πρέπει να προωθηθούν ώστε να, μπορούν να αξιοποιηθούν οι νέες επιγραμμικές υπηρεσίες και η πρόσβαση μαζί με τις νέες τεχνολογικές λύσεις προσφέροντας όλους τους Ευρωπαίους ασχέτως αν είναι ηλικιωμένοι, νέοι ή ε, με αναπηρίες. Όπως προείπα, σε ό,τι αφορά τις πλατφόρμες, αυτό ε, ε, ενδιαφέρει ιδιαίτερα στους σοσιαλιστές και δημοκράτες για να πλήξουμε τα μονοπόλια και τις δομές τους που θεωρούνται αθέμητα και άδικα για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Η προστεθέμενη αξία θα πρέπει να ε, είναι σαφής σε όλη την δομή της αλυσίδας παραχής υπηρεσιών. Για τις τηλεπικοινωνίες και την ευρυζωνική διακυβέρνηση και δομή είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ξεκάθαρου κανόνες με δίκαιο ανταγωνισμό και όπου υπάρχουν αποτυχίες στην αγορά θα πρέπει να συντομότερα τα διαθέσιμα μέσα, καθώς και τα ευρωπαϊκά κονδύλια, τι κρατικές βοήθειες και τις ε, επιτόπιες πρωτοβουλίες για το ευρωπαϊκό φάσμα, ώστε να ε, ε, τα εξοπλίσουμε όλα αυτά. Για την ψηφιοποίηση επίση, πρέπει να δούμε ποια είναι τα επόμενα βήματα που θα στηρίξουμε ω κοινοβούλιο. Θα πρέπει επίσης να εξασφαλίσουμε ένα υψηλό επίπεδο ασφάλεια στον κυβερνοχώρο με τους απαραίτητους κανόνες και το σχετικό κλάδο ως κλάδο προτεραιότητας. Είναι προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα στην ψηφιακή εποχή να έχουμε την ε, τυποποίηση των τεχνολογιών 5G οι πολίτες, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να έχουν εύκολη και απλή πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες. Επίσης, η Επιτροπή θα πρέπει να ολοκληρώσει την ανάλυση της προσεκτικά για το πώς η ψηφιοποίηση αλλάζει τις κοινωνίες μας και την καθημερινή μας ζωή. Οι Ευρωπαίοι πολίτες και οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν την απαραίτητη προστασία ε, και τα δικαιώματα τους να διασφαλίζονται και στον κυβερνοχώρο, ώστε να υπάρχει κοινωνική συνοχή και να προστατεύονται οι ευάλωτες ομάδες. Αυτά είναι ε, σημεία μία σημασία και δεν θα πρέπει να τα μιλήσουμε. Αυτή είναι η θέση που είχα να παρουσιάσω εξ ονόματος της ε, εισηγήτριας Μία Πέτερ. Ευχαριστώ. Η κυρία Φόρντ τώρα. Από πλευράς του ECR και συνεργασία και με τον άλλο σκιώδη του ECR. Θα ήθελα η έκθεση να στοχεύει, να επιτύχει ωφέλη και για τους καταναλωτές και για τις επιχειρήσεις να στηρίξει την καινοτομία και κάθε προσπάθεια ούτως ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας και να μπορέσουμε να αποφεληθούμε από την ψηφιακή ε, επανάσταση. Ευχαριστώ λοιπόν για την εργασία όλων. Να αναφερθώ σε μερικούς συμβιβασμούς πολύ συγκεκριμένα για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Δεν θέλω να είναι διαφορετικά τα δικαιώματα των καταναλωτών για το ίδιο απτό αγαθό. Αυτό ή το τηλέφωνό μου ή την τηλεόρασή μου. Ένα συγκεκριμένο καταναλωτικό αγαθό που να εξαρτώνται δηλαδή από τα αν τα αγοράζετε στο ίντερνετ ή από ένα κατάστημα. Αδιαφορεί ο καταναλωτής. Μπορεί να μπει σε ένα κατάστημα και να αγοράσει μια τηλεόραση ή να την αγοράσει στο διαδίκτυο. Όλοι λοιπόν οι σκιώδεις και οι συγκητές είμαστε όλοι σύμφωνοι ότι δεν πρέπει να υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση και αυτό λέμε στην Κομισιόν, παρακαλώ ακούστε μας, να το λάβετε υπόψη σας στο πώς προτίθεστε να έχετε άλλους κανόνες και άλλα δικαιώματα εάν οι αγορές γίνονται επιγραμμικά. Δεν συμφωνεί από αυτού το Κοινοβούλιο. Για το σύμβολο εμπιστοσύνης δεν θα ήθελα να υπάρχει ένα ενιαίο ενωσιακό επίπεδο να προκύψει από κάτω, από τους εμπλεκόμενους φορείς. Βεβαίως να εφαρμοστεί σωστά το άρθρο 20 της οδηγίας για τις υπηρεσίες για να μην υπάρχουν διακρίσεις. Σε όλη την ψηφιακή ενιαία αγορά θα έπρεπε να αξιοποιήσουμε όπου είναι δυνατόν την υπάρχουσα τοπολογία. Για το φάσμα. Δεν είμαστε υπέρ ενός εναρμονισμένου φάσματος Προσπαθήσαμε δύο φορές στο Συμβούλιο να το περάσουμε, δεν πάει. Άρα να υπάρχει συντονισμένη αντιμετώπιση του φάσματος για να επιτύχουμε πρόοδο. Να μην μπλοκάρει το θέμα και πάλι στο Συμβούλιο. Όλοι συμφωνούμε ότι δεν θέλουμε να υπάρχει ένας ε, και μοναδικός ε, ρυθμιστής για τις τηλεπικοινωνίες. Υπάρχει η BEREC, Πρέπει επίσης να ε, χρησιμοποιήσουμε καλύτερα και την ε, γλώσσα για το να ανοιχτεί η επιστήμη ακριβώς για να συντονίζεται με τον ορίζοντα 2020. Για τα ταχυδρομικά πακέτα δεν χρειάζεται να υπάρξει απόφαση από τα πάνω. Υπάρχουν προβλήματα σε ολισμενα κρατη κράτη-μέλη λειτουργεί και δεν είμαι υπέρ η Κομισιόν να έρθει σε άμεση επαφή με ε, τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας των κρατών μελών γιατί είναι κρατική αρμοδιότητα. Οι πλατφόρμες, οι καταναλωτές τις χρησιμοποιούν γιατί τους βολεύει. Πρέπει να έχουν αυτή την δυνατότητα. Είναι σημαντική λοιπόν η περιορισμένη ευθύνη των ενδιαμέσων. Αλλά βεβαίως πρέπει να έχουμε και τη φροντίδα για το καλό του καταναλωτή. Δεν συμφωνώ επίσης να επεκτείνουμε ε, με λανθάνοντα τρόπο την ε, την αρμοδιότητά μας και για θέματα κοινωνικής ασφάλισης. Επίσης, η κρυπτογράφηση είναι πολύ σημαντική και να λάβουμε υπόψη και την οδηγία Νίς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Επιτροπή Ήτρε, εκπρόσωπος ε, από πλευράς ε, ECR, ο κύριος Χένκελ. Οκ, okay, θα μιλήσω εγώ λιγότερο γιατί μίλησε πολύ η Βίκη. θα ασχοληθώ με τις παραγράφους 19 και 19α. Γιατί όλοι θέλουμε να υπάρχει ε, ευρυζωνικότητα και ε, γραμμές ε, υψηλής απόδοσης ακόμη και σε περιοχές της υπαίθρου. Και αυτό μπορούμε να το επιτύχουμε μέσω περισσότερου ανταγωνισμού και όχι λιγότερο. Δεν μπορούμε λοιπόν να αποδεχθούμε ολιγοπόλια για να επιτύχουμε επενδύσει. Αυτό είναι εντελώ λάθο. Σε σχέση με τις Ηνωμένε Πολιτείες, στην Ευρώπη, έχουμε προβλήματα γιατί φιλελευθερωποιήσαμε και ιδιωτικοποιήσαμε πολύ μετά τις Ηνωμένε Πολιτείε και ακόμη καθυστερούμε, υστερούμε έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν θα μπορέσουμε να καλύψουμε αυτή την καθυστέρηση εύκολα. Θα μπορούσαμε λοιπόν να προτείνουμε σε ορισμένες χώρες να πουλήσουν τις μετοχές που έχουν σε αυτούς τους φορείς οι δημόσιες αρχές. Ευχαριστώ. Το ECR συνολικά κράτησε το χρόνο του, περίπου. Η κυρία Ντίτα Χαράντζοβα από την Άλντε και από πλευράς Ίμκο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους συζητητές, τις για την προσπάθειά τους σε αυτό το δύσκολο θέμα. Συμφωνώ με την ε, άποψη της ΣΥΜΚΟ ότι πρέπει να έχει θετικό τόνο η έκθεση επιπλέον. Οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις αναμένουν να τους δώσουμε ε, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα ουσιώδη αποτελέσματα. Γι' αυτό η πολιτική ομάδα δεν συμφωνεί με τον συμβασμό για την παράγραφο, στην παράγραφο 7 ε, μέχρι και 11 γιατί ο συμβασμός αυτός πηγαίνει προς την αντίθετη κατεύθυνση. Φαίνεται ότι μερικές πολιτικές ομάδες θεωρούν ότι δεν πρέπει να αξιοποιήσουμε την ε, θετική προδιάθεση που ήδη υπάρχει για την ψηφιακή ενιαία αγορά και ότι δεν πρέπει να επιτύχουμε ενιαίους κανόνες. Στην ουσία πιέζουμε την Επιτροπή να καθυστερήσει για να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει για αυτό το 10% δοσοληψιών στο ίντερνετ. Να σας πω τι θα γίνει. Θα έχουμε 28 διαφορετικούς εθνικούς νόμους. Δηλαδή την τρέχουσα κατάσταση. Δεν είναι σωστό αυτό πιστεύω. Πρέπει να δράξουμε αυτή την ευκαιρία. Και εξάλλου δεν ισχύει ότι μια πρόταση που καλύπτει τις επιγραμμικές αγορές αγαθών και υπηρεσιών θα δημιουργήσει νομικό κενό μεταξύ αυτών των ε, αγορών και των άλλων αγορών. Γιατί αυτό το κενό ήδη υπάρχει. Η πρόταση της Κομισιόν θα ήταν ένα πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Και το δεύτερο βήμα θα ήταν αμέσως μετά, μόλις τελειώσει η διαδικασία Griffith. Νομίζω όμως ότι υπάρχει ακόμη δυνατότητα να καταλήξουμε σε αποδεκτό συμβιβασμό. πρέπει να αξιοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση τις αρμοδιότητές της όταν έχει, αλλά φυσικά δεν θα πρέπει να ασχολείται με θέματα για τα οποία δεν έχει αρμοδιότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε καμία από τις δύο επιτροπές μας. Γι' αυτό δεν μπορώ να δεχθώ πολλούς συμβαστικούς, ε, ε, πολλές προτάσεις συμβιβασμών των σοσιαλιστών, ιδιαίτερα για το τμήμα 3 δεν είναι θέμα δικό μας να μιλήσουμε για την κοινωνική ασφάλιση, για τα φορολογικά θέματα, για τα θέματα των δικαιωμάτων των εργαζομένων και του εργασιακού δικαίου. Βεβαίως έχουμε τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης. Αυτοί θα αποφασίσουν τι πρέπει να συμπεριληφθεί. Δεν πρέπει να μπει λοιπόν στους συμβιβασμούς μας. Και τονίζω ότι δεν είμαι επίσης υπέρ σήματος τεθέν της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα site στο ίντερνετ. Γιατί ξέρετε νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο για οποιοδήποτε να κάνει copy-paste ένα τέτοιο σήμα από ένα άλλο site στο δικό του. Ευχαριστώ κυρία μου, λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία Γιούλια Ρέντα από τους Πρασίνους και εκ μέρους της ΙΜΚΟ. Ευχαριστώ πολύ πρώτα απ' όλα τις εισηγητρίες και όλους τους κοιόδης που έχουν συμβάλει ως τώρα. Νομίζω ότι έχουμε προχωρήσει πολύ, ιδίως ε, στο θέμα ε, των πλατφορμών. Εάν κάνουμε διάκριση από τη μια από τις υποδομές, μεταξύ των υποδομών από τη μία και από την άλλη των υπηρεσιών, όπως είπε η κυρία Γκέπχαρτ, πολλά προβλήματα από αυτά που έχουν απομείνει μπορεί να αυτοεπιληθούν σε κάποιο βαθμό. Ίσως το θέμα της ουδετερότητας. Είναι σαφές ότι οι υποδομές πρέπει να είναι ουδέτερες, ενώ οι υπηρεσίες πολύ συχνά έχουν τη λειτουργία του φιλτραρίσματος. Έτσι λειτουργούν, δίνουν κάποια καθοδήγηση στους ε, χρήστες για τις ε, τόσες, ε, για τη σωρία πληροφοριών που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Πρέπει όμως να εξασφαλίσουμε την ουδετερότητα στις υποδομές. Επίσης, ακρό σημαντικό, να μην αποκλίνουμε από τη Γενική Αρχή της Οδηγίας Ηλεκτρονικού Εμπορίου για την περιορισμένη ευθύνη, διότι αυτό ήταν η βάση για τις υπηρεσίες του διαδικτύου που μπόρεσαν να ανθίσουν. Επίσης, ακούω τις μέρημνες, σημαίνω τις μέρημνες του ΕΛΚ για τις ροές ε, εισοδημάτων ε, και αντιτίμων για το περιεχόμενο ε, που διατίθεται από τους παρόχους. Θα πρέπει να δούμε τι μπορούν να αποκομίσουν ως αντίτιμο και τι κανόνε ισχύουν και για το ΦΠΑ λόγου χάρη, για τα βιβλία. Η πώληση στο διαδίκτυο καταλήγει σε υψηλότερη τιμή. Όμω τα ηλεκτρονικά βιβλία πολλούνται ω υπηρεσίε και όχι ω αγαθά. Το αν αλλάξουμε αυτό θα καθορίσει το κατά πόσο θα επιληθούν κάποια από τα θέματα προστασία καταναλωτή ω προ την πώληση ηλεκτρονικού περιεχομένου. Κατά αυτόν τον τρόπο λοιπόν νομίζω ότι μπορούμε να πετύχουμε ισόρροπα αποτελέσματα χωρί να θίξουμε τι υποκείμενε αρχέ του πώ αντιμετωπίζουμε την ευθύνη στο διαδίκτυο. Ε, Επίση, για να χτίσουμε μια οικονομία βασισμένη στα δεδομένα. Είμαστε σε καλό δρόμο συνολικά, όμως να ε, υποσημειώσω μια τροπολογία που έχουμε υποβάλει για την οδηγία ε, περιβάσεων δεδομένων. Είναι σημαντικό να μην ξεπεράσουμε εκείνα τα όρια, διότι έχουμε τώρα ένα νομοθέτημα όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ίδια έχει συμπεράνει ότι ε, έχει, δημιουργήσει, έχει λειτουργήσει ω τροχοπέδι στην ανάπτυξη της ηλεκτρονική οικονομίας. Εάν είμαστε σαφείς ότι θέλουμε την ηλεκτρονική διευθέτηση από τις αρχές της δεκαετίας του 90 ε, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η οδηγία αυτή είναι απερχιωμένη. Εάν θέλουμε οικονομία λοιπόν βασισμένη στα δόμενα στην Ευρώπη να την ξεφορτωθούμε. Και θα χρειαστούμε και στήριξη για τις προτάσεις μας για τις ανοιχτές επιστήμες και το σαφές πλαίσιο για την ε, ε, άγκληση δεδομένων είναι όλα αυτά σοβαρά ζητήματα αν θέλουμε η Ευρώπη να είναι ανταγωνιστική σε αυτό το τομέα και αν θέλουμε οι ερευνητέ μα να είναι σε θέση τα πορίσματά τους να τα διαθέτουν στο σύνολο της κοινωνίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία μου. Ο κύριος Ράιμον από την Ήτρε για τους Πρασίνους. Ευχαριστώ να ξανατονίσω τη σημασία του διαδικτύου και της ε, ψηφιακής αγοράς ως αρχοκοκαλιά της ε, κοινωνίας μας σίγουρα για την επόμενη δεκαετία και μάλλον και παραπάνω διότι ο τρόπος που θα την διαμορφώσουμε πρέπει να ε, λάβει αυτό το στοιχείο υπόψη. Πρέπει να μας απασχολήσει περισσότερο τι αντίκτυπος θα υπάρχει στην κοινωνία ε, πέραν από το απλό κέρδος λόγου χάρη να μην ξεχνάμε το θέμα του γεωγραφικού εντοπισμού ή αποκλεισμού. Ε, η πρώτη πρόταση ήταν πολύ καλύτερη από τη συμβαστική που, στην οποία καταλήξαμε και θα πρέπει να πιέσουμε, να πάψει ο γεωγραφικός αποκλεισμός. Αυτό μακροπρόθεσμα πρέπει να γίνει υποχρεωτικό. Θα πρέπει πρόσβαση σε κάθε σημείο και σε κάθε χώρα να είναι ελεύθερη. Η πρόσβαση στα δεδομένα να είναι απλή, εύκολη και χωρίς δυσκολίες. Επίσης να αναφερθώ σε δύο άλλα ζητήματα που επηρεάζουν ιδιαίτερα στην κοινωνία. Πρώτον, η ανάληψη πρωτοβουλίας από τις γυναίκες θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις τροπολογίες της συναδέλφου και από την Επιτροπή Γυναικών διότι η ψηφιακή οικονομία και τεχνολογία μπορεί να τους δώσει τεράστια μόχλευση στην ε, ε, πρόοδό του ω προ τα δικαιώματά του και αυτό θα πρέπει να αντικατοπιστεί και εδώ. Και για του ανθρώπου με αναπηρίε. Θα πρέπει και αυτό να απηχείται, διότι θα πρέπει λύσει να προσφερθούν όχι μόνον ε, ως προς τις εταιρείες που θα αρπάξουν ευκαιρίες στην αγορά, αλλά ευκαιρίες να έχει δικαίωμα να αντλήσει ολόκληρη η κοινωνία. Αυτές τις, ε, αυτό θέλουμε να επιτύχουμε τις δικές μας ε, προτάσεις για τις συμβαστικές λύσεις. Πιστεύουμε ότι η έκθεση συνολικά οδεύει κάπως την λάθος κατεύθυνση από την δική μας τη Σκοπιά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Για τώρα, δύο συνάδελφοι από την EFTD. Ο κύριος Μάρκο Τζούλο από την Επιτροπή ΙΜΚΟ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να συγχαρώ τις δύο εισηγήτριες για την δουλειά του. διότι ήταν περίπλοκο να βρούμε ένα σωστό σημείο ισορροπία μεταξύ των διαφορών τοποθετήσεων. Ώστε να μην υπάρξει υποβάθμιση, αλλά ε, να έχουμε ανωδική πορεία. Να επισημάνω ότι αυτή τη στιγμή ε, θέλω να επαναλάβω μια έκκληση που είχα ξανακάνει. Ε, ως προς την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη. Αυτό είναι ένας πυλώνας ε, στο χώρο του διαδικτύου. Νομίζω ότι η λειτουργία της ενιαίας αγοράς θα πρέπει για να είναι αποτελεσματική να βασίζεται στην εμπιστοσύνη. Το κείμενο λοιπόν αυτό που τώρα διατυπώνουμε πρέπει να δείχνει στον πολίτη ότι μπορεί να αισθάνεται ασφάλεια, εμπιστοσύνη. Ε, ακόμη και αν υπάρχουν καλά μέσα και εργαλεία στη διάθεσή του, ε, Εάν δεν αισθάνεται ασφάλεια και εμπιστοσύνη, δεν θα τα χρησιμοποιεί αυτά τα μέσα και εργαλεία. Δεν θα τα χρησιμοποιούνται όσα διατίθενται. Και πρέπει να φροντίσουμε αυτά τα εργαλεία να χρησιμοποιούνται. Ο πολίτη λοιπόν πρέπει κατά πρώτον να γνωρίζει, να έχει αντίληψη. Πρέπει να έχει μια συνολική εικόνα όλων των μέσων που έχει στη διάθεσή του. Κατά αυτόν τον τρόπο, εφόσον αποκτήσει αυτή τη συνολική εικόνα, θα κρίνει και αν είναι αποτελεσματικοί ή όχι οι κανόνε μα, οι προδιαγραφέ μα. Αυτή την εκκλήση την απευθύνω διότι περάσαμε από τι κατακαιρματισμένε τροπολογίε και τι διάφορε άσχετε ασύνδετε μνήε σε μια παράγραφο που μπορεί να κάνει συγκεκριμένη αναφορά και να μετουσιώνει αυτή τη συγκεκριμένη αίσθηση σε κάτι πιο χειροπιαστό. Ε, Ελπίζω να γίνει κάτι ακόμη πιο ε, ενταγμένο στο σώμα του κειμένου, ώστε αυτή η έννοια, αυτή η θεωρητική σκέψη να λάβει σάρκα και οστά. Πέρα από τα μέσα λοιπόν, εγγύηση ή οτιδήποτε άλλο, θα επαναλάβω ότι πρέπει να βρούμε ένα τρόπο να διατυπωθεί διαφορετικά ο κατάλογος των χειροπιαστών ενιών που θα ε, επιτρέπουν να δημιουργείται αυτή η σχέση εμπιστοσύνης ώστε να συμβούν όλα τα υπόλοιπα που θέλουμε να επιτύχουμε. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφε. Ο κύριος Μπορέλη, εκ μέρους της ΙΤΡΕ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και εγώ ε, ως συνεισηγητής. Ξέρω πόσο κοπιώδης ήταν η συμφωνία μεταξύ των διαφορών πολιτικών ομάδων. Ε, γι' αυτό συγχαίρω τις ε, συνεισηγητρίες Κάλλας και Κέπχαρτ για τη δουλειά τους. Πράγματι ήταν πολύ δύσκολο αυτό που προσπάθησαν, ιδίω ε, ω προ την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφόρων κοινοβουλευτικών επιτροπών. Ήταν ακόμη πιο περίπλοκο έτσι το έργο του. Ως ομάδα EFTD ε θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να συμβάλλουμε στην σύνταξη μιας έκθεσης που θα είναι ως το δυνατόν πιο ανοιχτόμυαλη, ε, εύληπτη, διεξοδική και ε, σε κάθε περίπτωση αισιόδοξη. Είμαστε πεπισμένοι ότι για να ολοκληρωθεί η νέα ψηφιακή αγορά θα πρέπει κεντρικό ρόλο να λάβουν οι πολίτες. Οπότε η ψηφιακή πολιτική δράση, η συμμετοχή των πολιτών είναι σημεία θεμελιώδου σημασία για μα. Άλλε πτυχέ, εξίσου σημαντικέ για μα, όπως τα γνωρίζετε αυτή εξ αρχής, είναι οι επενδύσεις στι υποδομέ. Για να διασφαλίσουμε την πρόσβαση στο βιζονικό φάσμα όλων και των οικογενειών ε, που μειονεκτούν και των ε, πολιτών στην Υπεθρό και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να δημιουργηθούν και νέε επιχειρηματικέ ευκαιρίε και νέε θέσει εργασία για όσου θέλουν να μπορούν να επενδύσουν ε, στον ψηφιακό χώρο. Σήμερα, μόνο το 14% της ευρωπαϊκής, του ευρωπαϊκού επιχειρηματικού κόσμου χρησιμοποιεί το διαδίκτυο ω βασικό διάβλο. Θα πρέπει λοιπόν οι δυνατότητε του ηλεκτρονικού εμπορίου να αξιοποιηθούν πλήρω. Είναι το νέο ε, όριο που θα έχουν να ξεπεράσουν στο μέλλον οι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Κάποιε μνήε στην ε, έκθεση υπάρχουν, το σημειώνουμε αυτό, αλλά κατά την άποψή μα θα μπορούσε να ε, αφιερωθεί ένα ειδικό κεφάλαιο της έκθεσης σε όλα αυτά. Επίσης η στατική σημασία της ε, ολοκλήρωσης της ψηφιακής αγοράς για την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο ώστε να δημιουργηθούν και να καινοτόμες θέσεις εργασίας. Θα πρέπει λοιπόν σε αυτή τη φάση να κάνουμε μια ε, υπέρτατη προσπάθεια να απογειωθούμε και η έκθεσή μας να είναι στο δυνατόν πιο φιλόδοξη. Να ε, κοιτάξουμε οι συμβαστικές μας προτάσεις να μην είναι τόσο ε, στραμμένες προς το πεζό ε, ε προς τον ορίζοντα χαμηλά, αλλά να κοιτάξουμε πώς θα μπορέσουμε να πετάξουμε. Πρόεδρος. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να μπορέσουμε να είμαστε στο τέλος όσο πιο ικανοποιημένοι γίνεται. Η κυρία Κάπελ. Ευχαριστώ. Και εγώ να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τους δύο συνεισηγητές, τις δύο συνεισηγήτριες για την πολύ καλή εργασία τους και για την ικανότητά τους να συνοψίσουν ένα τόσο περίπλοκο θέμα σε 38 συμβαστικές τροπολογίες αλλά και να κατανοήσουν το θέμα ευρύτερα και να επιτύχουν τόσο πολλούς συμβιβασμούς. Βεβαίως συμφωνούμε σε μεγάλο βαθμό ότι η ψηφιακή αλλαγή πρέπει να γίνει μέσω ενός ε, κανονιστικού πλαισίου ούτως ώστε να υπάρχει δίκαιος ανταγωνισμός για τις επιχειρήσεις και προστασία των καταναλωτών για να αξιοποιήσουμε το δυναμικό ανάπτυξης που έχει περιγράψει η Κομισιόν σε πολλές εκθέσεις και πολλές δημοσιεύσεις και για να επιτύχουμε και αύξηση της απασχόλησης. Πολλά ζητήματα είναι ανοιχτά, είμαι σίγουρη ότι θα διευκρινιστούν σύντομα από την πλευρά μας. Θέλω να τονίσω τρία σημεία. Παράγραφος 19 για τις ιδιωτικές ε, και δημόσιες ε, επενδύσεις 19-19α. Ε, ένας συνδυασμός των παραγράφων 19 και 20 για το εάν πρέπει εκ των προτέρων να ρυθμίζονται τα ολιγοπόλια, ιδιαίτερα στα πλαίσια της ανθεώρησης της οδηγίας για τις επικοινωνίες και ιδιαίτερα μας ενδιαφέρει το θέμα της ε, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Μας ενδιαφέρει να μην υπάρχουν διακρίσεις και ιδιαίτερα να μην γίνονται διακρίσεις σε βάρος των πιο ευάλωτων καταναλωτών. Επίσης τώρα η ιδιωτική χρηματοδότηση των υποδομών είναι πολύ σημαντικό να διατηρηθεί ο ανταγωνισμός γιατί αυτός ο καλύτερος τρόπος για να γίνουν επενδύσεις στις υποδομές. Αυτή τη στιγμή είναι ιδιαίτερα κρατικίστικο το κείμενο και δεν δημιουργεί ένα φιλικό πλαίσιο για επενδύσεις. Θα έπρεπε λοιπόν να τονίσετε ότι ο ανταγωνισμό για επενδύσει και για ε, ανάπτυξη υποδομών είναι θετικός. Δεύτερον, τα ολιγοπόλια. Κατά την άποψή μας, δεν είναι επιθυμητά για κανένα κλάδο της οικονομίας και αυτός ο κανονισμός εξάντε όπως προβλέπεται για την αγορά τηλεπικοινωνιών θα σήμαινε τρομερό βάρος για τις επιχειρήσεις και θα δημιουργούσε νομική ανασφάλεια. και αυτό πρέπει να το συζητήσουμε και στα πλαίσια της αναθεώρησης για τις τηλεπικοινωνίες, του πλαισίου της τηλεπικοινωνίες. Ιδιαίτερα πρέπει να θέσουμε το θέμα της ε, συνδεσιμότητας και να καλύψουμε τα κενά στα πλαίσια της επόμενης γενιάς προϊόντων. Είναι σημαντικό να ελέγξουμε λοιπόν να λειτουργεί αυτό το ρυθμιστικό πλαίσιο και να δημιουργήσουμε ενάυσματα για να αναπτυχθούν περισσότερο τα δίκτυα. Και τέλος, ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Βεβαίως, Πρέπει οι γυρεότεροι καταναλωτές, οι καταναλωτές στην Ήπεθρο να έχουν ε, εύκολη πρόσβαση, αλλά να μην υφίστανται διακρίσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για την ε, πολύ καλή αυτή συζήτηση. Η κυρία Βίκη Φόρντ θα προεδρεύσει για το υπόλοιπο της συνεδρίασης. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ πολύ, θα σας πω τον κατάλογο των ομιλητών. Olga Shinalova, Zander, Lisa Yakansari, Gunnar Hotmark, Dan Dalton, Antonis Claire Moody, and then the Commission. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξέχασα κανέναν? Παρακαλώ σηκώστε το χέρι. Μάικλ, ναι, εσείς είσαι στον κατάλογο. Ο Μάικλ θα είναι ο πρώτος ε, γιατί ήταν ο συντάκτης γνωμοδότησης στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Έχει το λόγο λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις ε, συνεισηγήτριες αυτής της έκθεσης για την εξαιρετική δουλειά τους και ελπίζω ότι θα ολοκληρώσουμε την εργασία αυτή την επόμενη εβδομάδα. Να σας ενημερώσω επίσης ότι εμείς εχθές ψηφίσαμε στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ ε, την δική μας συμβολή στην έκθεση αυτή και νομίζω ότι είναι μια ισορροπημένη ε, πρόταση παρουσιάζουμε την προστασία των δεδομένων από την άποψη των θεμελιωδών δικαιωμάτων, αλλά επίσης υπάρχει ισορροπία μεταξύ θεμελιωδών δικαιωμάτων και ε, ανάπτυξης των επιχειρήσεων, επεξεργασίας των δεδομένων, όπως επίσης και μία νέα άποψη για την ασφάλεια. Οπότε ελπίζω ότι η συμβολή μας θα είναι σημαντική ε, στη δική σας έκθεση και ελπίζω ότι θα τη μεταχειριστείτε με σοβαρότητα όταν ε, θα φτάσετε στην τελική εκδοχή της έκθεσής σας ε, καταλαβαίνετε, καταλαβαίνοντας και το, τη σημασία του άρθρου 54 και το τελευταίο μου σχόλιο είναι για τις πλατφόρμες. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να μην είμαστε πολύ περιοριστικοί, να λάβουμε υπόψη και το μέλλον, να μην είμαστε πολύ περιοριστικοί με πάρα πολλές μεθόδους, με πάρα πολλούς κανόνες για τις πλατφόρμες. Νομίζω ότι αν δεν κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση, θα είναι καλύτερος ο συμβιβασμός. Δεν χρειάζεται να ε, καταστρέψουμε τις ήδη υπάρχουσες πλατφόρμες. Ευχαριστώ. Ο Γιώσε Μπλάνκο. Α, Μπλάνκο Λόπε. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και του συζητητέ, τις συζητήτρες για την εργασία τους. Γιατί ένα θέμα τόσο περίπλοκο το αντιμετώπισαν πολύ σωστά. Πρώτον, ευχαριστώ τις αναφορές που γίνονται στην ε, προσπάθεια που πρέπει να γίνουν για να καλύψουμε το ε, ψηφιακό χάσμα. Είναι πολύ σημαντικό για όλους και για τους οργανισμούς αυτοδιοίκησης και για μένα που προέρχομαι από μια περιοχή που ζει προβλήματα έντονα γύρανσης και φτώχειας. Βεβαίως πρέπει να σταματήσει επίσης και ο αποκλεισμός ορισμένων γεωγραφικών περιοχών γιατί αυτό οδηγεί σε καταστάσεις ε, διακρίσεων. Δεν ξέρω ε, αν έχουμε παλαιότερη εκδοχή των ε, συμβαστικών 16 και 18. Στη 18 λέει ότι θα πρέπει να δούμε εάν οι περιορισμοί στην γεωγραφική πρόσβαση ε, παραβιάζουν τους όρους ανταγωνισμού και είναι διακρίσεις ε, με βάση τον ε, πάροχο υπηρεσιών του καθενός. Αλλά δεν είναι δυνατόν να δικαιολογείται ο γεωγραφικός αποκλεισμός. Και δεύτερον, ο περιορισμός με βάση τη διεύθυνση του παρόχου επιγραμμικών υπηρεσιών οφείλεται στο ότι ορισμένα στοιχεία του περιεχομένου ε, έχουν εγκριθεί μόνο για ορισμένε περιοχές. Στο 16 λένε ότι το μπλοκάρισμα αυτό, ο αποκλεισμό ορισμένων γεωγραφικών περιοχών ενθαρρύνει την πειρατική ε, χρήση περιεχομένου. Αυτό είναι λάθος. Αυτό που ευνοεί την ε, πειρατική χρήση περιεχομένου είναι ότι δεν εφαρμόζονται οι προδιαγραφές το γεγονός ότι κάποιοι μπορούν να δούνε ταινίε, για παράδειγμα που έχουν δικαιώματα είναι το βασικό. Νομίζω ότι με τέτοια λογική θα έχουμε περιορισμούς αδικαιολόγητους. Πρέπει λοιπόν να ξαναδούμε την ε, σύνταξη αυτών των δύο συμβασμών. Ευχαριστώ πολύ. η Όλγα Συναλόβα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τις ε, ε, συνεισηγήτριες και τους συμπροέδρους. Θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια για τις συμβιβαστικές τροπολογίες. Πρώτο σχόλιο αφορά την πρόσβαση για όλους τους πολίτες. Νομίζω εδώ δεν θα έπρεπε να μας διαφεύγει ότι πολλοί πολίτες, κυρίως πιο ηλικιωμένοι, οι οποίοι δεν είναι ή δεν μπορούν να είναι τμήμα της ε, ηλεκτρονική κοινωνία, παρά το γεγονός ότι εγώ είμαι υπέρ βέβαια τη καθολική πρόσβασης όλων των πολιτών και της ε, πλήρους ε, ένταξης στην ε, ψηφιακή κοινωνία δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσουμε να παρέχουμε υπηρεσίες στον πραγματικό κόσμο. Για παράδειγμα, τη δυνατότητα να πάει κάποιος σε ένα γιατρό για να πάρει μία συνταγή. Νομίζω ότι αυτή η δυνατότητα πρέπει να διατηρηθεί και να αναφέρεται αυτό και στην έκθεση. Δεύτερο σχόλιο αφορά την παράγραφο 16 που αφορά το ε, geo-blocking. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει μία άνηση πρόσβαση λόγω της γεωγραφικής θέσης και αυτό είναι κάτι που δεν αφορά μόνο τον ψηφιακό κόσμο αλλά και τον πραγματικό κόσμο και νομίζω ότι και η Επίτροπος Γιώροβα το είχε παραδεχθεί αυτό όταν είχε έρθει στην Επιτροπή μας. Οι κανόνες και για τον κόσμο του διαδικτύου αλλά και για τον πραγματικό κόσμο πρέπει να είναι κανόν, να είναι ίδιοι, να μην κάνουμε διακρίσεις υπέρ του ενός ή του άλλου και γι' αυτό η πρόσβαση με βάση τη γεωγραφική θέση δεν θα έπρεπε να ξεφεύγει από τον κανόν αυτό. Εγώ ήμουν μία από τις σκιώδεις εισηγήτριες για την Επιτροπή Μεταφορών. Νομίζω ότι η γνωμοδότησή μας είναι πολύ καλή η οποία θα, και θα έπρεπε να ενσωματωθεί στη δική σας δουλειά. Έχουμε συμπεριλάβει πολλές πτυχές και θα χαρούμε ιδιαίτερο αν κάποια από τη συμβολή μας ε, ενσωματωθεί στην ε, μελλοντική δική σας δουλειά. Σας ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Από την Επιτροπή Ιτρε Αν Σάντερ. Όχι. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ζήτησα το λόγο, αλλά άμα μου το δίνετε το λόγο, ευχαρίστως ε, να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία. Σας ευχαριστώ πολύ. Δύο λόγια θα πω. Να ευχαριστήσω και εγώ ε, τις συνεισηγήτριες για τη δουλειά τους ε, και κυρίως για όσα πρόκειται να κάνουν θα ήθελα να πω ότι εγώ είμαι μέλος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και με την ιδιότητά μου αυτή νομίζω ότι είναι σημαντικό να διατηρηθούν δύο ιδέες. Πρώτον, ότι η ψηφιακή ενιαία αγορά μπορεί να παρέχει κάποιες ευκαιρίες ε, σε μισθωτούς που δεν θα τις είχαν ε, ε, διαφορετικά και αναφέρομαι κυρίως για όσους βρίσκονται στις περιοχές της υπαίθρου, βέβαια η διατύπωσή μα στην Επιτροπή απασχόληση είναι πολύ ευρύτερη και γι' αυτό είναι αναγκαίο να εκπαιδεύσουμε τους ανθρώπους αυτούς και να τους δώσουμε τις απαραίτητες ικανότητες. Να επιμείνω σε ένα δεύτερο σημείο, το οποίο ε, αφορά περισσότερο την δική σας επιτροπή και αναφέρομαι στις πλατφόρμες. Μου άρεσε αυτό που είπε ο κύριος Ζουβέν για την ευθύνη, για την ευθύνη των πλατφορμών και αναφέρομαι κυρίως στη δυνατότητα ανάληψης ε, ε, δέσμευσης ε, για πελάτες που είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και που δεν μπορούν να υπερασπιστούν πάντοτε τον εαυτό τους, να μπορέσουμε δηλαδή να τις μεταχειριστούμε με πιο δίκαιο και διαφανή τρόπο. Αυτές λοιπόν ήταν οι ιδέες που θα ήθελα να εκφράσω εγώ διαβάζω όσους βρίσκονται στον κατάλογό μου. Antinas Gorgas and Claire Moody. Would anybody else like to signal for the floor? No? Okay. Θέλει κάποιος άλλος το λόγο? Όχι, ευχαριστώ. Η κυρία Γιακονσάρη δεν είναι εδώ, οπότε ο Γκούναρ Χουέκμαρκ. Ευχαριστώ, Οπότε θα πάρω το, την ώρα και της ε, συναδέλφου. Να ευχαριστήσω κατά πρώτον τις δύο που Πολύ δύσκολη δουλειά σας. Και ως ο πρόεδρος ο Γερζη Μπούζεκ Μα επέτρεψε να δούμε το θέμα ξανά και ξανά, διότι ήταν δύσκολο να είμαστε ικανοποιημένοι. Ε, αλλά, Πρόεδρε, νομίζω ότι είναι λάθος να λέμε ότι δεν θα καταλήξουμε όλοι να είμαστε ικανοποιημένοι. Πρέπει να γίνει αυτό. Ε, και να έχουμε ένα μεγάλο επίπεδο φιλοδοξιών. Θα ζήσουμε σε ψηφιοποιημένο κόσμο, θέλουμε δεν θέλουμε. Η ερώτηση είναι αν θέλουμε να έχουμε πενταχωριστικό ρόλο ή όχι. Μια σκέψη για τις συμβαστικές ε, λύσεις, χωρίς να μπω σε λεπτομέρειες, μπορώ να κάνω γενικώ. Ε, μια παρατήρηση. Θα πρέπει πιο πολύ να μετριάσουμε τις συνέπειες σε μια αλλαγή που έτσι κι θα γίνει, παρά να περιορίσουμε τις ευκαιρίες. Νομίζω ότι είμαστε μία από τις μεγαλύτερες οικονομίες στον κόσμο, ιδίω ε, ψηφιακού χαρακτήρα. Κανείς δεν θα υποφεληθεί όσο εμείς. Γι' αυτό να είμαστε βέβαιοι ότι θα έχουμε πρωταγωνιστικό ρόλο. Πρώτα απ' όλα στο 5G. Στο 5G θα έχουμε ε, την τυποποίηση ουσιαστικά του διαδικτύου. Η ψηφιοποίηση ήταν ένα, ένα βήμα, το 3G, το 3G δηλαδή ήταν ένα άλλο. Το 5G θα είναι ένα τεράστιο βήμα. Αν δεν αναδράξουμε αυτή την ευκαιρία ώστε να ε, ορίσουμε το τι θα γίνει με το φάσμα, την νομοθεσία περί ΦΠΑ, ώστε να μετατραπούμε σε ψηφιακή οικονομία, με τα ηλεκτρονικά βιβλία λόγου χάρη, εάν υπερρυθμίσουμε τις πλατφόρμες που διαρκώς μεταλλάσσονται, θα περιορίσουμε τις ευκαιρίες και θα ήθελα να ζητήσω από τους συνεισηγητές κατά κάποιο τρόπο να διαψεύσουν τον Γέρζη σε αυτό που είπε ξανά και ξανά. Ότι ε, ο στόχος είναι να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Εάν δεν μπορέσουμε να θέσουμε τον πύχη πολύ ψηλά και να έχουμε ένα μεγάλο ύψος προσδοκιών, άλλοι θα ε, καταλάβουν την πρώτη θέση. Θα μείνουμε δεύτερη και τρίτη, για να μην πω και τέταρτη. Δεν θα μας αρέσει, ούτε θέλω να βρεθούμε σε αυτή τη θέση. Δεν θα μου αρέσει κάτι τέτοιο γέννηση. Ε, νομίζω ότι ο στόχος μας είναι να είμαστε πρώτοι. Τότε θα ήμασταν όλοι ευχαριστημένοι, πιστεύω. Πολύ ωραία. Πρώτη, πρώτη. Ο κύριος ε, Ντάλτον. Ευχαριστώ τι συνεισηγητριέ γιατί κάνατε πολύ καλή δουλειά λόγω του μεγάλου αριθμού τροπολογιών και των πόσων συναδέλφων συμμετείχαν στην όλη δουλειά. Ε, δεν είμαι ικανοποιημένο με όλα. Νομίζω δεν θα πρέπει να αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά περισσότερο η οι φορεί στην αγορά για τα σήματα εμπιστοσύνη, για το γεωγραφικό αποκλεισμό, νομίζω ότι πρέπει να κοιτάζουμε και πώ σχετίζεται αυτό με το περιεχόμενο και αν κάτι δεν διατίθεται σε ένα συγκεκριμένο κράτο μέλο, να το δούμε επιμέρου. Δεν ξέρω αν ε, τεχνικώ είναι δυνατό αυτό. Πάντω η δική μα συνεδρία σηματοδοτείται μέσα από το διαδίκτυο σε τον κόσμο. Τίποτα ε, εμπόδιο δεν υπάρχει εδώ. Οπότε ο στόχο είναι να υπάρχει ω το δυνατόν πρόσβαση. Για το cloud computing, το υπολογιστικό νέφο, εδώ πρέπει να παραμένουμε κοντά στι παγκόσμιε εξελίξει και να μην ακολουθήσουμε αυτή την προσέγγιση που τώρα υπάρχει, είναι λάθο για τα ε, δικαιώματα των καταναλωτών. Έχω πραγματικέ ανησυχίε για την δικαιωτική μεταχείριση, για τι υπηρεσίε που είναι διαθέσιμε στο διαδίκτυο ή όχι, την σωστή διάκριση για το φάσμα. Ε, να πω ότι ναι, χρειάζεται βελτιωμένο συντονισμό, αλλά όχι αναδομονισμένη πολιτική φάσματο. Αυτό είναι ένα θέμα επικουρικότητα κατά μένα. Οπότε συνολικά, παρά την πολύ καλή δουλειά, λείπει νομίζω το κεντρικό νόημα. Αυτό που τώρα είπε και ο Γκούναρ Χέκμαρτ. Εδώ ο στόχο δεν είναι να διαθετήσουμε τα πράγματα για του καταναλωτέ του διαδικτύου. Ε, ακολουθούμε μια παλαιομοδίτικη προσέγγιση. Ε, δεν μα ενδιαφέρει εδώ να διατυπώσουμε ένα δόγμα και να μα έχει ξεπεράσει το μεταξύ ο κόσμο, ούτε μπορούμε να ξαναβάλουμε το τζίνι πίσω στο λιχνάρι. Ε, δεν υπάρχει τρόπο να γίνει αυτό. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και να αποσπάσουμε τα ωφέλη τη ψηφιακή οικονομία. Όχι όπως τώρα, γιατί αυτό δεν θα μας βοηθήσει για τους στόχους μας στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπόγκα. Ευχαριστώ. Είναι συναπαστικό το θέμα και χαίρομαι πολύ που είμαι πιο κοντά σήμερα στους σοσιαλιστές και δημοκράτες, αλλά είναι ένα πολύ ωραίο κοκτέιλ αυτό που έχει γίνει σοσιαλιστών και φιλελευθέρων. Πραγματικά σας εύχομαι λοιπόν κάθε καλή τύχη για να ε, πετύχει το θέμα αυτό και η εξέταση του. Νομίζω με την εμπειρία της Γερμανίας μπορείτε να προσφέρετε πολλά, διότι εάν δεν πετύχει ε, η έκθεση αυτή, δεν θα έχουμε πολλές ευκαιρίες ως Ευρώπη. Και εδώ ε, υποκρύπτονται πολλές ευκαιρίες για τους νέους. Ε, όλοι έχουν να κερδίσουν από αυτό το, από την ψηφιακή οικονομία, από το διαδίκτυο. Όλοι στην Ευρώπη εδώ έχουμε μια τεράστια ευκαιρία και χρειαζόμαστε λοιπόν ισχυρότερη διατύπωση που να δείχνει ότι η Ευρώπη είναι ανοιχτή στην κοινοτομία και μία ε, οικονομία που να επιτρέπει την ε, σωστή κατανομή. Ε, οι πλατφόρμες είναι το μέλλον, οι πλατφόρμες υπάρχουν, οι άνθρωποι είναι εξετρελαμένοι με τις πλατφόρμες, μα αφήστε τους να το ευχαριστηθούν και να λειτουργήσουν όπως θέλουν οι πλατφόρμες. Τι δείχνει το DSM. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι γίνεται με τις ε, ταχυδρομικές υπηρεσίες, τις ε, παραδόσεις δεμάτων και τις αγορές. Εδώ υπάρχουν δυσκολίες. Αφήστε τις επιχειρήσεις να πουλάνε, αφήστε το να προχωρήσει, αφήστε το να εξελιχθεί. Δεν, μαρε, δεν με ενδιαφέρουν τα σήματα εμπιστοσύνη, ούτε αυτό ενδιαφέρει τους, τον κόσμο, τους ψηφοφόρους μας. Οπότε ας μην ε, επικεντρωθούμε σε αυτό. Δεν είναι τόσο σημαντικό. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να μπορούν να λειτουργήσουν ε, ελεύθερα όλα στο διαδίκτυο. Όσο περισσότερους φραγμούς προβλέψουμε, τόσο μεγαλύτερες δυσκολίες δημιουργούμε. Ας το επιτρέψουμε λοιπόν όλο αυτό να πραγματοθεί. Ας βεβαιωθούμε ότι όλοι μπορούν να ωφεληθούν. Η Κλέρ Μούντι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τις συζητήτριες και τους κοιόδης για το Ηράκλειο έργο που έχουν επιτελέσει. Και όλοι ελπίζουμε ότι θα επιτύχουμε όλους τους συμβασμούς που επιδιώκουμε για τον συμβασμό 22α και αυτά που λέτε για τον Μπέρεκ και ότι πρέπει να έχει την επαρκή χρηματοδότηση που του αρμόζει. Βεβαίως, το καλωσορίζω. σε σχέση με ορισμένα που άκουσα. Οπωσδήποτε πρέπει να αναγνωρίσουμε πόσο ευρεία είναι η ψηφιακή ενιαία αγορά. Δεν αφορά τους πολίτες μόνο ως καταναλωτές, τους αφορά και ως πολίτες γενικότερα. Αυτό αφορά το Συμβασμό 19α, όπου τονίζεται την αναγκαιότητα να γίνουν επενδύσεις για καθολική πρόσβαση στην ευρυζωνικότητα και πρόσβαση στην ψηφιακή ενιαία αγορά. Αλλά και ευρύτερα μας ενδιαφέρει να μην αποκλείεται κανείς από την ψηφιακή οικονομία. <coughs> να μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση σε δεξιότητες. Όχι μόνο μέσω της παραδοσιακής κατάρτισης σχολείου πανεπιστήμιο, αλλά σε όλη τη διάρκεια του εργασιακού του βίου. Να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης όλων. Να μην υπάρχουν αποκλεισμοί. Αυτό σημαίνει και πρόσβαση σε εργασιακά δικαιώματα. Γιατί η ψηφιακή οικονομία πρέπει να επιτρέπει στους πολίτες να εργάζονται. Αλλά όταν εργάζονται πρέπει να έχουν την ίδια προστασία που θα είχαν εάν ε, εργάζονταν διαφορετικά. Και πρέπει να θεωρούν δεδομένη αυτή την προστασία. Σόλ Κέλλερ. Οι τελευταίοι τέσσερις ομιλητές ήταν πιο λογικοί. Πολύ καιρό έχω να ακούσω τόσο λογικά πράγματα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Και νομίζω ότι ο Γκούναρ ήταν ο πρώτος που μίλησε σωστά λέγοντας ότι ναι, μπορούμε να δώσουμε χαρά στους ανθρώπους. Και δεν θα πρέπει να υπάρχει αντίφαση μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων. Αν είναι ευτυχεί οι επιχειρήσει, θα είναι ευτυχεί και οι καταναλωτέ. Αν προστατεύουμε τα άτομα, διευκολύνουμε και την ανάπτυξη που θα ε, βοηθήσει τα άτομα. όσοι συγητής ε, Ήτρε ασχολούμαι με τον κανονισμό για τα δεδομένα και την προστασία δεδομένων και κοντεύουμε να καταλήξουμε. Και ο τριμερής διάλογος ελπίζω να λήξει πριν τα Χριστούγεννα. Σήμερα έκανα μία ερώτηση για την έρευνα και ρώτησα οι ερευνητέ είναι ικανοποιημένοι γιατί αν δεν μπορούν να δουλέψουν με αυτό το πλαίσιο τότε δεν επιτύχουμε τους στόχους μας 3% του ΑΕΠ για την έρευνα και φυσικά η έρευνα ε, ωφελεί και τους καταναλωτές. Αυτά λοιπόν που ο Γκούνερ και ο κύριος Ντόλσον και οι υπόλοιποι, όλα αυτά είναι πολύ σωστά σημεία, πρέπει να συμπεριληφθούν στο κείμενό μας ούτως ώστε ο κανονισμός αυτός να διατηρήσει την Ευρώπη στην, στην πρωτοπορία. Θέλουμε να είμαστε στην πρώτη θέση, όχι στη δεύτερη. Και μπορούμε να το επιτύχουμε. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα να δώσω το λόγο στην Επιτροπή. Και μετά στους ε, δύο συνσηγητές. Αλλά έχουμε και λίγο περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας. Αν κάποιος κοιόδης ε, θέλει να προσθέσει κάτι, μπορούν, ε, μπορεί να μου το πει τώρα. Μήπως η Επιτροπή θέλει να μας πει τίποτα. Ο κύριος Ντεγάρ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχω ένα γενικό σχόλιο και δύο ειδικά. Το γενικό είναι ότι καλωσορίζουμε τη μνήμα στη συμβαστική τροπολογία για το κοινό σύνολο κανόνων διότι το πρόβλημα της ψηφικής αγοράς είναι ότι έχουμε κατακαιρματισμό 28 διαφορετικά σύνολα κανόνων. Εάν θέλουμε ενιαία ψηφιακή αγορά πρέπει να έχουμε μία αγορά και ένα σύνολο κανονα προφανώς. Αυτό απαιτεί μία άλλη διαδικασία νομοθέτησης και εδώ και στο Συμβούλιο. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η ελάχιστη εναρμόνιση δεν είναι ο τρόπος να οδεύσουμε προς μία νέα ψηφιακή αγορά. Δεν μπορούμε να έχουμε 28 συν ε, ένα σύνολα κανόνων. Θα πρέπει τα 28 να αθρηστούν και να γίνουν ένα. Θα βεβαίως να δούμε τι θα γίνει και στην ε, πράξη. Οπότε και την πρώτη δοκιμασία θα την έχουμε σύντομα. Αυτόν τον ε, στόχο θα τον γνωρίζουμε πολύ γρήγορα, αν θα, γνωρίζουμε πολύ γρήγορα πρόβλημα να επιδιώξουμε. Θέλουμε ταχύτητα. Θα δούμε ε, λοιπόν πώς θα πάνε τα πράγματα στην αγορά. Η νομοθεσία πρέπει να προχωρήσει γρηγορότερα και η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα είναι πολύ στοχευμένη, ώστε και οι συνομοθέτες να μπορέσουν να δράσουν άμεσα. Δύο συγκεκριμένες παρατηρήσεις για το γεωγραφικό αποκλεισμό. Νομίζω από τις συμβαστικές τροπολογίες φαίνεται το Κοινοβούλιο να πιστεύει ότι μπορούμε να ξεφορτωθούμε το γεωγραφικό αποκλεισμό με καλύτερη υλοποίηση του άρθρου 20 της Οδηγίας για τις Υπηρεσίες και με το δίκαιο ανταγωνισμού ε, ιδίω με τα όσα προβλέπονται από το ηλεκτρονικό εμπόριο και τη σχετική οδηγία. Εμείς ε, καταλήξαμε ότι χρειαζόμαστε νομοθετικά μέτρα για να ξεφορτωθούμε τον γεωγραφικό αποκλεισμό. Χρειάζεται η εφαρμογή του άρθρου 20. Είναι και επιθυμητό και απαραίτητο αυτό. Αλλά είναι απαραίτητη προπόθεση, όχι όμω είναι ικανή είναι αναγκαία, αλλά όχι ικανή προπόθεση. Δεν θα επιληθεί έτσι το πρόβλημα του γεωγραφικού αποκλεισμού. Γι' αυτό ε, ε, καλωσορίζουμε την στήριξη του Κοινοβουλίου προς αυτήν την κατεύθυνση. Με την έκθεση που ετοιμάζεται δεν έχετε ε, ε, δεν έχετε εκφραστεί για την νομοθετική ανάγκη να επιληθεί έτσι το, ε, ο γεωγραφικό αποκλεισμό. επίση για τα τηλεοπτικοακουστικά, τα πνευματικά δικαιώματα τοποθετήθηκαν κάποιοι ε, βουλευτές, τα αγαθά που κάποιοι αγοράζουν στο διαδίκτυο και εκεί υπάρχουν περιπτώσεις γεωγραφικού που θα παρατηρήσει για τις πλατφόρμες. Θέλουμε να αποφύγουμε την εντύπωση ότι κάτι ε, υπάρχει εκεί έξω που το ονομάζουμε έτσι θεωρητικά πλατφόρμες. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με τις πλατφόρμες. Διότι εάν δούμε τις ε, περιοχές όπου προχωρεί γρήγορα η κοινοτική νομοθεσία, το θέμα των πλατφορμών παντού εμφανίζεται. Τηλεπικοινωνίες, ισότιμοι κανόνες, οπτικοακουστικά, ε, πνευματικά δικαιώματα, το ανέφεραν κάποιοι ε, βουλευτέ στο ψηφιακό χάσμα, γεωγραφικό αποκλεισμό, ασφάλεια στον χώρο. Παντού συζητιέται το θέμα που αφορά τι πλατφόρμες. Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε τι δράση χρειάζεται, αλλά να αποφύγουμε την εντύπωση <laughs> ότι οι πλατφόρμε δεν μπορούν να διαθετηθούν ή δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη καθώ κοιτάζουμε σημαντικά νομοθετήματα ε, και πώς ε, πρέπει να επικυροποιηθούν για να λειτουργήσει η ενιαία ψηφιακή αγορά. Εάν μου επιτρέπετε, πριν επανέλθω στους ε, εισηγητές, όταν φτάσουμε στην ψηφοφορία, οι, οι γνωμοδοτήσεις των επιτροπών που έχουν ε, γνωμοδοτήσει θα συμπεριληφθούν στον κατάλογο ψηφοφοριών. Και επίσης επεξεργαζόμαστε και τον κανονισμό για την προστασία των δεδομένων ταυτόχρονα στο Κοινοβουλίο. Υπάρχει το θέμα της ασφάλειας ε, των πληροφοριών και η σχετική νομοθεσία. Ε, είναι σκιώδης εισηγητής εδώ ο Γέρζη. Θα πρέπει εδώ να φροντίσουμε να συμπορεύονται αυτά που προβλέπουμε εδώ για την ασφαλεία στον χώρο. Διότι ελπίζω ότι θα ολοκληρωθούν, θα φτάσουν σε πέραση δύο περίπου ταυτόχρονα. Οπότε καλό θα είναι να δούμε τα δύο ζητήματα από κοινού. για να είμαστε και σαφείς και εύστοχοι στο ότι ψηφίζουμε στις 14. Οι δύο εισηγήτρες τώρα, κυρία Κεπχάρτ, εσείς πρώτη ή κυρία Κάλλας. Κυρία Κάλλας. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και για τα σχόλιά σας. Μερικά ζητήματα στα οποία ήθελα να σταθώ Έχουμε σε πολλές περιπτώσεις το πρόβλημα ότι κανείς δεν βλέπει την συνολική ευρωπαϊκή εικόνα και έχουμε 28 διαφορετικά σύνολα κανόνων. Θα πρέπει να ε, παρακολουθεί κάποιος ε, συνολικά την ευρωπαϊκή εικόνα, όμως ε, πρέπει με τη διατύπωσή μας να ενισχύσουμε το ρόλο του Μπέρεκ. Δεν θα πρέπει να προβλέψουμε έναν νέο οργανισμό. Για τις ε, πλατφόρμες λυπούμε που ο κύριος Ζουβά έχει φύγει από την αίθουσα, αλλά όπως είπε θέλουμε να είμαστε μεν πρώτοι ε, στην ψηφιακή οικονομία, αλλά αυτό που θα πρέπει να έχουμε κατά νου είναι ότι οι πλατφόρμες ως ε, διάμεση έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία της ψηφιακής οικονομίας και προκειμένου αυτή να αναδυθεί. Εάν λοιπόν προβλέψουμε μεγαλύτερες ευθύνες για τους ενδιάμεσους, ίσως οδηγήσουμε σε συρρήκνωση την ψηφιακή οικονομία, γιατί επιτρέπουμε στους ενδιάμεσους να παρέχουν υπηρεσίες, και αν έχουν ε, σοβαρότερε υποχρεώσει, αυτό σημαίνει ότι ε, λιγότερε εταιρείε θα δραστηριοποιούνται στην αγορά. Αυτό ε, πιστεύω ότι είναι κάτι σημαντικό. Πρέπει να το κατανοήσουμε. Και επίση, κάτι άλλο πρέπει να έχουμε κατά νου είναι ότι οι πλατφόρμες δεν έχουν να κάνουν μόνο με το πολιτιστικό περιεχόμενο. Υπάρχουν και άλλε πλατφόρμε πολύ διαφορετικού είδου. Είναι φοβερή επικοινωνία. Επίσης, θα πρέπει να δούμε και το καθήκον ε, ε, και τη διάκριση από την ευθύνη. Οι πλατφόρμες ε, τείνουν να αποφεύγουν τον κίνδυνο, το ρίσκο και γι' αυτό υπάρχουν λιγότερε εταιρείε στην αγορά. Ω προ την πρόσβαση για όλου υπάρχουν σχετικέ παράγραφοι, οπότε συμφωνώ απολύτω ότι τα ζητήματα αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη. Και για την φορητότητα, όπω αυτό είναι αρμοδιότητα τη Επιτροπή ε, Νομικών Υποθέσεων, θα περιμένουμε και τη δική του γνωμοδότηση αλλά συμφωνούμε απολύτως. Το περιεχόμενο που έχει αγοραστεί θα πρέπει να μπορεί να μετατοπίζεται για το γεωγραφικό αποκλεισμό. Από τη μια ήταν αρμοδιότητα της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων, από την άλλη μα ζητήθηκε να συμπληρώσουμε το πλαίσιο για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Δηλαδή, ο γεωγραφικός αποκλεισμός και οι σχετικές πρακτικές όταν δεν είναι δικαιολογημένες θα πρέπει να πάψουν. Νομίζω λοιπόν συμφωνούμε επί των περισσότερων παρατηρήσεων και θα συμφωνήσω απολύτω με αυτά που υπόθηκαν για τη θετική προσέγγιση ε, σχετικά με τις ευκαιρίες που, που προσφέρει η ψηφιακή οικονομία. Θα πρέπει να το τονίσουμε αυτό και όχι να μιλούμε μόνο για τους κινδύνους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Γκέπχαρτ. Ο κύριος Μπούζεκ δεν μπορεί να μείνει πολύ ακόμη. Γιατί σε δύο ώρες πρέπει να πάει σε δεξίωση ενώπιση των Χριστουγέννων. Κυρία Γκέπχαρτ. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομη. Θα προσπαθήσω τουλάχιστον. Καταρχάς, το καθήκον μας δεν είναι οι πολίτες, οι βουλευτές να είναι ευτυχείς ο καθένας πρέπει να βρει μόνος του την ευτυχία. Γιατί για τον καθένα είναι κάτι διαφορετικό η ευτυχία. Είναι διαφορετικό αυτό που τον χαροποιεί και αυτό που τον λυπεί. Δεν είναι νομίζω μια συζήτηση που πρέπει να κάνουμε. Αυτό που είναι ουσιώδες είναι να είμαστε απόλυτα σαφείς. Η καινοτομία της ψηφιακής αγοράς μας δίνει τρομερές ευκαιρίες και πρέπει να τις αδράξουμε. Σαφές αυτό. Αυτές τις ευκαιρίες σχετίζονται με το οικονομικό μας μέλλον και θέλουμε να είμαστε πρωτοπόροι, αριθμός ένα στον κόσμο. Αλλά να διευκρινίσω και κάτι ακόμη. Γιατί ξέρετε κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις. Η μία όψη είναι πάντα η θετική, η αντίστροφη είναι η κίνδυνη που συνδέονται και ως υπεύθυνη πολιτική δεν μπορούμε να πούμε θα τονίσουμε μόνο το θετικό. Όχι. Πρέπει να ασχοληθούμε και με το προβληματικό. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να λύνουμε αυτά τα προβλήματα που προκύπτουν. Παράδειγμα, για το θέμα που ανέφερε η κυρία Φόρτ, η παράγραφοι 7, 8 και 19α όπου λέμε ότι πρέπει να είναι ίδια η κατάσταση για το αν αγοράζει κανείς το ίντερνετ ή όχι το ίδιο προϊόν. Και συμφωνούμε σχεδόν όλοι σε αυτό. Και στις συμβαστικές τροπολογίες σχεδόν όλες οι πολιτικές ομάδες είπαν αυτό ακριβώς. Οι μόνοι που είναι κατά είναι οι φιλελεύθεροι. Όλοι οι άλλοι που εκφράστηκαν είπαν σαφώς αυτό που θέλουμε είναι να ισχύουν τα ίδια για τις αγορές στο ίντερνετ και εκτός. Άρα τι άλλο μπορούμε να βάλουμε συμβαστικές. Αυτά που λένε οι περισσότεροι. Η προφανής πλειοψηφία όπως προέκυψε από τις συζητήσεις. Και γι' αυτό αυτά λένε και οι συμβαστικές τροπολογίες. Και λυπάμαι που οι φιλελεύθεροι ε, δεν συμφωνούν με τις παραγράφους 7 έως 11 και δεν θέλουν να συνυπογράψουν. Αλλά τι να κάνω, λυπάμαι, έτσι έχουν τα πράγματα. για τους συμβιβασμούς για τον γεωγραφικό ε, αποκλεισμό. Είναι πολύ δυσχερές θέμα, γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να κάνουμε μία διάκριση μεταξύ του γεωγραφικού αποκλεισμού για ορισμένα μέσα, όπως βίντεο, κινηματογράφος, τηλεόραση, και τον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, του επιγραμμικού εμπορίου, που είναι κάτι διαφορετικό. Πρέπει να γίνει αυτή η διάκριση. Και γι' αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σε διαφορετικά σημεία για να διευκρινίσουμε ότι πρέπει να ισχύουν ενδεχομένως διαφορετικές διατάξεις. Γιατί όταν αγοράζω μια τηλεόραση δεν ασχολούμαι τόσο πολύ με πνευματικά δικαιώματα όσο όταν αγοράζω ένα βίντεο. Είναι σαφές αυτό. Πρέπει να γίνουν λοιπόν οι κατάλληλες διακρίσεις. Αλλά δεν πρέπει να γίνεται διάκριση αν αγοράζει κανείς το ίδιο προϊόν επιγραμμικό σημείο. Περί αυτού πρόκειται. Για το άρθρο 20, οδηγία για τις υπηρεσίες. Μπορεί να μας βοηθήσει σε πολλούς τομείς, αλλά όχι σε όλους. Πρέπει να λάβουμε υπόψη πολύ πιο συγκεκριμένα και το δίκαιο ανταγωνισμού που μπορεί να μας βοηθήσει ιδιαίτερα για τις κανονιστικές διατάξεις για τις πλατφόρμες σε σχέση με την ιδιαιτερότητα του δικτύου σε συνδυασμό δηλαδή με αυτό, για να έχουν όλοι τις ίδιες ευκαιρίες. Οι μικρές επιχειρήσεις, οι start-up που ξεκινάνε, να έχουν την ίδια δυνατότητα να συμμετάσχουν στις πλατφόρμες όπως και οι μεγάλες που είναι ήδη εκατεστημένες και έχουν ε, τη θέση τους. Αυτά πρέπει να τα δούμε. Δεν μπορούμε να τα παραβλέψουμε. Βεβαίως θέλουμε πρόοδο, αλλά επίσης πρέπει να δούμε Πώς θα βοηθήσουμε, πώς θα δώσουμε τις ίδιες ευκαιρίες στις μικρομεσαίες και τις νέες επιχειρήσεις. Αυτό πρέπει να εξετάσουμε. Για ποια σημεία προκύπτουν προβλήματα και άρα χρειάζονται λύσεις. Βεβαίω, μα ενδιαφέρουν και όλα όσα υπόθηκαν για την πρόσβαση για τα άτομα με αναπηρίες. Και αυτά πρέπει να μας απασχολήσουν, γιατί είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Και θα μας απασχολήσουν και ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ε, πολλές πολύ καλές προτάσεις που υπευλήθησαν από, τη, από τις διάφορες επιτροπές και ελπίζω να τα καταφέρουμε να διατυπώσουμε και τους τελευταίους συμβασμούς να είναι τόσο καλοί όσο οι προηγούμενοι έχουμε εργαστεί πολύ, θα συνεχίσουμε να εργαζόμεθα και νομίζω, νομίζω ότι τελικά θα είναι πολύ καλό το κείμενό μας ακόμη και αν ε, ο καθένας μας θα μπορούσε να πει «Αχ, αν το είχα γράψει μόνος μου θα ήταν πολύ διαφορετικό», αλλά και αυτό φυσιολογικό. Αλλά ε, μέχρι στιγμής είμαι πολύ ευχαριστημένη από τη συνεργασία μεταξύ όλων ε, των ομάδων και αυτά που ήδη έχουν επιτευχθεί, τουλάχιστον η δική μου ομάδα τα υποστηρίζει μέσω μου. Ευχαριστώ πολύ. λαμπρά. Ευχαριστώ όλους όσους άκουσαν τη συζήτηση αυτή. Ξέρω ότι θα ενσωματωθεί στη διαδικασία συμβιβασμού. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο σε αυτός ο συμβιβασμός. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους ε, τους βοηθούς μου, τη γραμματεία. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Πολλές λεπτομέρειες ε, για τις οποίες ακόμη πρέπει να συμφωνήσουμε. Θα ήθελα να είμαι πρακτική και να σας υπενθυμίσω ότι ψηφίζουμε στις 14 Δεκεμβρίου, Δευτέρα βράδυ στο Στρασβούργο. Και ξέρω ότι μερικές φορές κάποιοι συνάδελφοι φτάνουν αργά, έπτα η ώρα το βράδυ θα γίνει η ψηφοφορία. Παρακαλώ πολύ να το κανονίσετε έτσι ώστε να είστε παρόντες 7 η ώρα το βράδυ. Δεν ξέρω αν κανείς θέλει να το συζητήσει αυτό. Ο κύριος Κέλλη, κάθε φορά που έχουμε ψηφίσει ε, Δευτέρα βράδυ στην Ολομέλεια είναι 9 η ώρα το βράδυ. Γιατί αυτή τη φορά είναι 7. Πολλοί κόσμος ταξιδεύει εκείνη την ώρα και από τη Φραγκφούρτη όταν έρχεται κανείς ε, μπορεί να είναι πάρα πολύ δύσκολο λόγω ε, της κίνησης. Ναι, μπορούμε να το συζητήσουμε και να προσπαθήσουμε να ψηφίσουμε αργότερα, αλλά πρέπει να το συζητήσουμε με τους συντονιστές. Γνωρίζω ότι κάποιες επιτροπές όταν ε, ψηφίζουν Δευτέρα βράδυ αρχίζουν λίγο πιο αργά, αλλά τότε ε, πάει πολύ αργά η συνεδρίαση. Φτάνουμε δηλαδή μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Ε, ίσως θα μπορούσαμε να αρχίσουμε 8.30 λέει ο κύριος Μπούζεκ ή 8 η ώρα μέχρι τα μεσάνυχτα. Θα συμφωνήσουμε μέσω των συντονιστών, αλλά να σας πω, αγαπητοί συνάδελφοι, πολύ σημαντική παρατήρηση. Είναι σημαντικό ο Κίνερ Χόκμαρκ ενδεχομένως να μπέρδεψε δύο πολύ σημαντικούς όρους. Δυστυχώς εξαφανίστηκε. Δεν μπορώ να του το εξηγήσω λοιπόν του ιδίου. Πολύ φιλόδοξο ε, όταν κάτι είναι πολύ φιλόδοξο δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει συμβιβασμός. Εγώ δεν είπα να μην είμαστε όσο το δυνατόν πιο φιλόδοξοι για τους καταναλωτές μας ε, προκειμένου να οικοδομήσουμε τη σωστή αγορά για τους πολίτες αλλά και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για τις ε, ψηφιακές επιχειρήσεις ο συμβιβασμός όμως είναι απαραίτητος αγαπητοί φίλοι, διαφορετικά δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε την εργασία μας. Απλώς μερικές φορές με το συμβιβασμό δεν μπορούμε να επιτύχουμε όλα όσα προσδοκούμε. Και μπορεί εν μέρη να είμαστε δυσαρεστημένοι. Να το επαναλάβω λοιπόν, μία ακόμη φορά, διαφορετικά δεν είμαστε έτοιμοι για συμβιβασμό. φιλόδοξο, το να είναι κάτι φιλόδοξο και το να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε συμβιβασμό είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Μπορούμε να είμαστε φιλόδοξοι, αλλά τελικά θα χρειαστεί ένα συμβιβασμό. Δυστυχώ. Η κυρία Φόρντ. Πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ψηφοφορία μέχρι τις 9 το βράδυ από ό,τι κατάλαβα. Τέλος πάντων θα επανέλθουμε για το θέμα της ώρας ψηφοφορίας. Έχουμε ήδη συμφωνήσει επί πολλών συμβιβαστικών τροπολογιών, οπότε ας είμαστε ικανοποιημένοι. Κάποια ζητήματα μπορεί να χρειαστεί να ψηφιστούν και γι' αυτό ακριβώς